πρόεδρος, είπε η πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Monday uh, Τη Δευτέρα το απόγευμα έρχονται σιγά σιγά όλοι έρχονται, αλλά τα υπόλοιπα ας τα πω γερμανικά. Την ημερήσια διάταξη την ελάβατε, η κυρία Βασιλείου η Επίτροπος δεν μπορεί να έρθει γιατί συνέβη, είχε ένα θάνατο στην οικογένεια και θα έρθει σε κάποια από τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Προσωπικά, <laughs> πολύ ευτυχής που δεν θα έρθει γιατί το Μάιο η Κομισιόν στη, θα μιλήσει για νέες προτάσεις. Οπότε αν έρθει το Μάιο θα ξέρει περισσότερα και θα έχει περισσότερο νόημα η συζήτηση, θα είναι πιο απτά τα θέματα. Συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Τώρα τα πρακτικά της περασμένης συνεδρίασης υπάρχει. Αν έχετε πρόβλημα κατά τη διάρκεια του απογεύματος να μας ενημερώσετε, αλλιώς το βράδυ θα θεωρηθούν και εγκριθέντα. Υπενθυμίζω ότι πάλι γίνεται τηλεοπτική αναμετάδοση της συνεδρίασης βαλτικές γλώσσες δεν έχουμε, ούτε μαλτέζικα, ούτε σουηδικά. Θα καλωσορίσω με μια νέα συνεργάτητα, την Φαμπιέν Κοντεβίλ, με τα μακριά μαύρα μαλλιά που πρόσφατα ήρθε στη γραμματεία μας και προέρχεται από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τώρα πέρασε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Καλή επιτυχία και καλή δουλειά. Όπως είπα ήδη, η Επίτροπος είναι ήδη εδώ. Είναι υπεύθυνη για ένα πολύ λεπτό θέμα, ένα φάκελο που συζητείται πολύ από εμάς. Ε, έχουμε την εισηγήτρια και τους σκιώδεις που ήρθαν ειδικά σήμερα για να συζητήσουν μαζί της. Οπωσδήποτε είναι σημαντικό να κάνουμε τις παρατηρήσεις για το πρόγραμμα της Κομισιόν θα της δώσω το λόγο να κάνει την εισαγωγή στις εργασίες της και σίγουρα θα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχετε τον λόγο κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόσκλησή σας. Και το θέμα δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε προαναγγείλει, αλλά θα ήθελα να κάνω πρώτα ένα ιστορικό των τελευταίων μηνών. Μέχρι και ένα χρόνο πριν. Θα γνωρίζετε ότι η δέσμη broadband είχε εγκριθεί το Σεπτέμβριο με τρία κύρια θέματα που τα γνωρίζετε από τη σχετική ανακοίνωση μαζί με την πολιτική για το Radio Spectrum Policy Program και την πρόσβαση της επομένης γενναίας Next Generation Access, τη σύσταση. Παρακολούθησα τι συζητούσατε κι εσείς στην Επιτροπή σας και τι εξηγούσατε στον έξω κόσμο και γνωρίζω τι φρονείτε. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Γιατί συμφωνούμε ότι είναι κάτι το σημαντικό και τα καταφέρατε θαυμάσια. Τώρα για το Radio Spectrum Policy Program. Δεν χρειάζεται νομίζω να σε εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να βρουν κάποιο πρακτικό τρόπο να προχωρήσουν ως προς την ουσία για να υπάρξει κάποια πρόοδο στην εφαρμογή των προτάσεων. Μπορεί να υπάρξουν ορισμένες δυσκολίες, αλλά θα τα καταφέρουμε μάλλον. Κατανοήσαμε πλήρως κυρία Πρόεδρε, όλα όσα έθιξε η Επιτροπή σας και θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι η Κομισιόν εκτιμά ιδιαίτερα τη σημασία των συχνοτήτων και του σπέκτρουμ για τον πολιτισμό και για τις εκπομπές. Να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις παρακαλώ. Όπως γνωρίζετε είμαι πραγματιστικός άνθρωπος και Πρέπει νομίζω να αποφύγουμε ιδεολογικές διαμάχες μεταξύ των διαφόρων ειδών μέσων μαζικής ενημέρωσης έτσι ώστε να παίξει η ευρεία πρόσβαση τον πλήρη ρόλο που πρέπει να παίξει. Γιατί είναι και αυτός ένας τρόπος ε, πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. Το δεύτερο, η δεύτερη νομοθετική δέσμη πέρυσι αφορούσε την κυβερνασφάλεια και ιδιαίτερα τον εξυγχρονισμό του ΕΝΙΣΑ. Πρόσφατα κάναμε την αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης 2009 και έγινε μια ανακοίνωση στις 31 Μαρτίου που θα συζητηθεί σε υπουργική διάσκεψη στην Ουγγαρία αυτή την εβδομάδα στις 14 και 15 Απριλίου. Τώρα σε αυτά που σας ενδιαφέρουν πιο άμεσα. Όπως ανακοινώθηκε κατά ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή σας τον περασμένο Νοέμβριο, η Επιτροπή Σοφών υπέβαλε την έκθεσή της η νέα αναγέννηση στην Επιτροπή στις 10 Ιανουαρίου και συμπεριλαμβάνει πολύτιμες συστάσεις για την πρόσβαση σε πολιτιστικό περιεχόμενο, στη ψηφιοποίηση και σε πρακτικές λύσεις για τον εξυγχρονισμό των πνευματικών δικαιωμάτων. Πράγμα που με φέρνει τώρα στο Ευρωπαϊκά. Η συλλογή αυτή έχει αυτή τη στιγμή 15 εκατομμύρια κομμάτια και ο αριθμός των επισκεπτών έχει τριπλασιαστεί. Η αριθμή αυτή είναι εντυπωσιακή γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τόσο σημαντικές επιτυχίες χωρίς να αγνοούμε πάντοτε τον τελικό στόχο βέβαια. Υπάρχουν και καινούργια σχέδια όμως. Η Επιτροπή σας θα έπρεπε να τα συζητήσει. Ίσως όχι σήμερα, αλλά άλλη φορά. Η γεωτάφτιση του περιεχομένου για εφαρμογές κινητών συσκευών, φορητών συσκευών που θα σας δείχνει πού βρίσκονται τα κοντινότερα στοιχεία στην Ευρωπιάνα. Υπάρχει το πρόγραμμα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που επιτρέπει στους πολίτες να έχουν εικόνες, γράμματα, κάρτ ποστάλ και άλλα αντικείμενα μέσα στα πλαίσια του, της Ευρωπαϊάνας. Άλλο θέμα που γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει και σας είναι η προστασία των ανηλίκων στο ίντερνετ. Και εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί τα παιδιά χρησιμοποιούν πολύ πιο πρόθυμα τις νέες τεχνολογίες τους αρέσει να μαθαίνουν καινούργια πράγματα όπως τα βίντεο και πρέπει τα παιδιά μας να έχουν και την πρόσβαση αλλά και την προστασία που αξίζουν οι υπηρεσίε μου προετοιμάσουν μια έκθεση για την εφαρμογή των συστάσεων 98 με 2006 για την προστασία των ανηλίκων και την δήλωση για τα βιντεοπαιχνίδια. Θα λαμβάνουν υπόψη τους και την ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και την ανάπτυξη των παιχνίων στο ίντερνετ. Η Επιτροπή λοιπόν συνεχίζει να παρακολουθεί την εφαρμογή του των αυτορυθμιστικών αρχών μας για ένα πιο ασφαλές κοινωνικό δίκτυο. Έγιναν βέβαια όλες οι διαβολεύσεις που απαιτούνταν με τους ενδιαφερόμενους και για την ουδετερότητα του δικτύου και για το roaming. Σε λίγο θα κάνουμε μία ανακοίνωση για την ουδετερότητα του δικτύου επιμένοντας σε, στον ανοιχτό του χαρακτήρα την καινοτομία και στη διαχείριση των υπηρεσιών και για το roaming θα κάνουμε πρόταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011. Για τη μεταφορά της νομοθεσίας οι δύο κυριότερες εξελίξεις είναι ο καθορισμός του Μπέρεκ και η διορία της 26ης Μαΐου για το πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών. Αν χρειαστεί θα κάνουμε και προσφυγές για παραλήψεις αν υπάρχει κάποιο κράτος που δεν εφαρμόζει τους κανόνες που πρέπει να εφαρμόζει. Η Κομισιόν θα επιμείνει για τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες όπως τα θέματα της χώρας προέλευσης και τα θέματα της δικαιοδοσίας που ισχύει καθώς και την προστασία των ανηλίκων και το δικαίωμα απάντησης. Τον προηγούμενο μήνα στείλαμε γράμματα σε 16 χώρες μέλη για να βεβαιωθούμε ότι η εφαρμογή της οδηγίας ε, γίνεται σωστά και μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερος γύρος επιστολών. Τρεις χώρες μέλη, Πολωνία, Πορτογαλία και Σλοβενία, ακόμη δεν μας έχουν γνωστοποιήσει τι συνοδευτικά μέτρα λαμβάνουν και μπορεί να γίνουν αντικείμενο προσφυγών. Άλλο τώρα προκλητικό και ενδιαφέρον θέμα, η έρευνα. Βρισκόμαστε στα μέσα της εφαρμογής του 7ου προγράμματος πλαισίου. Το 2011 είναι το σημαντικότερο έτος αυτού του προγράμματος με 1,2 δισεκατομμύρια που έχουν διατεθεί. Πέρα από τα 780 εκατομμύρια που είχαν διατεθεί από την διάσκεψη του Σεπτεμβρίου του 2010. Επίσης, αναλαμβάνουμε προγράμματα για να διευρυνθούν τα κοινωνικά ωφέλη όπως καλύτερη πρόσβαση στο δίκτυο και ενεργή και υγιής γύρανση. Τον περασμένο Νοέμβριο εδώ στο Κοινοβούλιο έγινε μια παρουσίαση των θετικών πτυχών της λεγόμενης προσβάσιμης ψηφιακής τηλεόρασης ώστε να μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητές της και τον Νοέμβριο με τον συνάδελφό μου Ιωάννη Ντάλη Επίσης ε, εγγενίασα το πρώτο πιλωτικό υπηρεματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα καινοτόμας εταιρικής σχέσης για την ενεργή και υγιή γύρανση που σκοπεύει μέχρι το 2020 να καταστήσει τους πολίτες ικανούς να ζουν περισσότερο με καλύτερη υγεία. Αυτό το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε συνεργασία με μας και τους ενδιαφερόμενους. Έτσι θα πλησιάσουμε περισσότερο σε μια βιώσιμη και πιο κοντά στους πολίτες ανάπτυξη. Επίσης υπάρχει το πρόγραμμα δράσης για την ήτακη διακυβέρνηση που ε, είχε υποβληθεί στις 15 Δεκεμβρίου 2010 για να μπορέσουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν πραγματικά την ενιαία αγορά εκμεταλλεύοντας τις δημόσιες υπηρεσίες και χρησιμοποιώντας πλήρως τις ηλεκτρονικές δημόσιες προμήθειες. Γενικότερα θα αρχίσουμε να ετοιμάζουμε ήδη τον διάδοχο του προγράμματος ε, πλαισίου 7, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο που θα συμπληρωθεί από την διάσκεψη του ψηφιακού προγράμματος 16 και 17 Ιουνίου εδώ στα Βρυξέλλας. Ελπίζω πολλοί από εσά να συμμετάσχουν γιατί θα είναι πολύ σημαντική διάσκεψη και ενδιαφέρουσα. Τώρα για τον δομημένο διάλογο. Τι μπορεί να αναλάβουμε το 2012 που είναι το έτος κλειδί για συγκεκριμένη δράση αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Και πρέπει να τους πετύχουμε πρόθεσμα, ζητώ την υποστήριξή σας για τις θετικές συστάσεις της Επιτροπής των Σοφών. Σε μερικούς έστειλα επιστολές από σας. Μπορεί τα ωφέλη για την κοινωνία μας να είναι να δεκαπλασιαστούν αν ψηφιοποιήσουμε τον πολιτισμό μας. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται βέβαια και πιο βαθύτερη συζήτηση και με εσάς όλοι μας και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και η Ευρωπαϊάνα έχουν σαφέστατους στόχους αλλά ίσως δεν καταφέραμε 100% να το εκφράσουμε με την διπλωματική γλώσσα που απαιτείται για να μπορεί ο κόσμος ευρύτερα να αναγνωρίσει τη σημασία της Ευρωπαϊάνας όπως θα έπρεπε για να την εκμεταλλευτεί πλήρως. Χρειάζεται να κάνουμε ακόμη πολλά λοιπόν παρά το ότι Ήδη έχουμε κάνει αρκετά. Μόνο όμως αν μπορέσουμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. Θα προτείνουμε λοιπόν ένα νέο πρότυπο χρηματοδότησης και υπάρχει και η αναθεώρηση της σύστασης του 2006 για την ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα πολιτιστικού υλικού και την ψηφιακή του διατήρηση. Επίσης θα θέλαμε να προωθήσουμε γενικότερα τις πληροφορίες που διαθέτει ο δημόσιος τομέας σε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο το 2012. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε και τα παραδείγματα που μπορούν να μας δώσουν τα κράτη-μέλη. Η Επιτροπή έχει τα πρώτα αποτελέσματα μιας μελέτης για το ψηφιακό πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Κληρονομιά δημόσια διαβούλευση θα ακολουθήσει και εργαστήρια και μπορεί να υποβάλουμε μέτρα για την κινηματογραφική κληρονομιά στην τρίτη μας έκθεση για την εφαρμογή του, της σύστασης για την κινηματογραφική κληρονομιά του 2005. Τον Ιούνιο του 2010 μας ζητήσατε να αξιολογήσουμε τις πολιτικές πτυχές του λεγόμενου Internet of Things διαδικτύου των πραγμάτων για να ωφεληθεί ακόμη περισσότερο η αγορά και οι πολίτες από αυτό. Πρόσφατα ανακοινώθηκε μία παγκόσμια συμφωνία για βελτίωση της πρόσβασης στις ραδιοφωνικές συχνότητες και την περασμένη εβδομάδα υπέγραψα μία εθελοντική συμφωνία με τη βιομηχανία, την κοινωνία των πολιτών, την Ενίσα και το ενωσια... τις ενωσιακές αρχές προστασίας δεδομένων ώστε να γίνουν προτάσεις για καλύτερη προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα των δεδομένων. Αυτό το πρόγραμμα πλαίσιο για την προστασία του ιδιωτικού χαρακτήρα των δεδομένων στις ραδιοφωνικές εφαρμογές είναι το πρώτο τέτοιο έγγραφο στην Ευρώπη. πρόκειται λοιπόν για ιστορική συνάντηση, πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί εκεί είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πράγμα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, συνήθως ο καθένας επιμένει στα δικά του. Τελικά όμως υπήρξε και κάποια συμφωνία, πολύ δύσκολα όλα αυτά και τελικά αποδείχτηκε μεγάλη επιτυχία η εκδήλωση αυτή και κανείς δεν έθεσε αντιρρήσεις. Επίσης εξετάζουμε την πιθανότητα να προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για την ενιαία αγορά που να αφορούν την ήττα ταυτότητα και τις ΙΤΑ υπογραφές για να υποστηρίξουμε έτσι την ενιαία αγοραστική πράξη ή ενιαία πράξη της αγοράς ή πράξη της ενιαίας αγοράς. Αυτά τα συστήματα θα καταστήσουν δυνατό για τους πολίτες να επωφεληθούν από τις δημόσιες υπηρεσίες που χορηγεί η ενιαία αγορά παντού σαν να βρισκόταν παντού στην δική τους χώρα. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε όταν μιλάμε για ενιαία αγορά στα ψηφιακά. Ότι τα σύνορά της δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν σύνορα. Και η τα ταυτότητα, η ήττα ταυτοποίηση, η ήττα υπογραφή είναι πράγματα που θα διευκολύνουν αυτή την κατάργηση των συνόρων. Όπως λέει λοιπόν το ψηφιακό πρόγραμμα, η Κομισιόν θέλει να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερα ωφέλη από το συνδυασμό της λειτουργίας των διαφόρων συστημάτων και εξετάζει την πιθανότητα να καθοριστεί ένας ελάχιστ, μια ελάχιστη κοινή δέσμη ε, δεδομένων ασθενών για να μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση έτσι ώστε να σώζονται περισσότερες ζωές. Το 2012 επίσης θα συμπληρωθεί η προσπάθειά μας για την ανάλυση και επεξεργασία ενός σχεδίου δράσης υπό την αιγίδα του προγράμματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Στρατηγική Υπολογισμού των Συνέφων ή των Νεφών. Πολλοί από εσάς. έχετε διασυνδέσεις αλλά δεν ξέρετε όλοι ότι το κοινό μας στοιχείο είναι ο πολιτισμός και οι κοινότητές μας και η ανοιχτή πρόσβαση και η ουδετερότητα του δικτύου οι ραδιοφωνικές εκπομπές δημοσίου χαρακτήρα η ήττα διακυβέρνηση, ο ιδιωτικός χαρακτήρας και φυσικά γενικότερα η ασφάλεια είναι κάτι που θα ρόλο τους, είναι πράγματα που θα παίξουν το ρόλο τους και αυτά. Πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη για να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και τώρα περιμένω τα δικά σας σχόλια. Γιατί εδώ παίζονται πολλά και υπάρχει και πίεση χρόνου. Πρέπει να είμαστε όλοι βέβαιοι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουμε τη συζήτηση λοιπόν, η οποία είναι ευρύτατη. Η κυρία Κάμα Εβερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για τις ε, παρατηρήσεις σας. Δεν θα σας εκπλήξει ότι επανέρχομαι στο Radio Spectrum Program λέτε ότι θέλετε να λειτουργήσετε πραγματιστικά σε αυτό το τομέα. Δεν νομίζω ότι άλλωστε είναι ιδεολογική αντιπαράθεση εδώ. Πρόκειται για διαφορετικά συμφέροντα που πρέπει να συγκεράσουμε με ισορροπημένο τρόπο. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Και στην Επιτροπή μας έχουμε συμφωνήσει ότι η βελτίωση της ευρείας ζώνης στην Ευρώπη έχει σχέση με την πρόσβαση στην επικοινωνία και στην πληροφορία. Πρέπει να τα εγγυηθούμε αυτά. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου το κλασικό ραδιόφωνο μακροπρόθεσμα χρειάζεται ακόμη σύνορα και γι' αυτό θέση στην Επιτροπή μας ήταν ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για ε, ένα ψηφιακό dividend 2 ενώ ξέρουμε ότι Ορισμένα κράτη-μέλη δεν έχουν αρχίσει ούτε το Digital Dividend 1 και γι' αυτό η προθεσμία για την εφαρμογή του 1 έχει παραταθεί μέχρι το 2015 και όσοι μπορούν θα τηρήσουν την αρχική ε, καταληκτική προθεσμία το 2013. Γι' αυτό λέμε πώς αρχίζουμε με το ψηφιακό κομμάτι 2 ενώ ξέρουμε ότι αυτά αφορούν πολύ το ραδιόφωνο και όχι μόνο τα κρατικά προγράμματα αλλά και την ιδιωτική ραδιοφωνία. Στη Γαλλία το 80% για παράδειγμα των τηλεοπτικών μεταδόσεων γίνονται μέσω επιγείων συστημάτων καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας. Ένας τομέας ο οποίος αποτελεί σημαντικό, ε, σημαντική συνιστόσα της ε, ελευθερίας των ΜΜΕ και της ενημέρωσης. Οπότε πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προστασίας τουλάχιστον ε, στο βαθμό που ξέρουμε ότι ακόμα ο τομέας χρειάζεται την προστασία. Και καλό θα ήταν, θα είμαστε ευγνώμονες, αν ως Επίτροπος λαμβάνατε υπόψη αυτή τη θέση το Radio Spectrum Program. Επίσης η ασύρματη ραδιοφωνία μας απασχολεί πολύ και ξέρουμε ότι πολλά κοινοτικά θέατρα δυσκολεύονται πολύ. Το έχουμε ζήσει στη Γερμανία διότι το γεγονός ότι δεν είχε διευκρινιστεί εκ των προτέρων ποιος θα είναι υπεύθυνος για τα αντισταθμιστικά μέτρα ε, ε, είχαμε προβλήματα και στη Γερμανία είχαμε με το Digital ε, Dividend 1 και αυτά μπορούν να επαναληφθούν και στην Ευρώπη. Οπότε εκ των προτέρων θα πρέπει στα κράτη-μέλη να διευκρινίζεται ποιος, πώς και σε τι ύψος θα υπάρχει αντιστάθμιση και αποζημίωση όταν ε, αλλάζουν οι συχνότητες και οι εκπομπές για να μην ε, επαναληφθούν τα προβλήματα της Γερμανίας όπου τώρα ξαφνικά κανείς δεν ε, θεωρεί αυτόν υπεύθυνο και τα θέατρα είναι μόνα τους, τα δημοτικά επίσης. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορούν να καλύψουν οικονομικά αυτά τα μέτρα. Καλό είναι λοιπόν εκ των προτέρων να προβλέψουμε τι ακριβώς θα γίνεται και πώς θα αντιμετωπίζονται τα νέα προβλήματα. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς σε ποιο βαθμό είστε διατεθειμένοι ως Επίτροπος να λάβετε υπόψη σας αυτά τα δύο θέματα που είναι κεντρική σημασία για την Επιτροπή Πολιτισμού στα πλαίσια του Radio Spectrum Program και να ε, διασφαλίσω με τη θέση των, ε, της κρατικής ραδιοφωνίας, αλλά βέβαια και τον, ε, τη χρήση ασύρματων μικροφώνων κλπ. Ευχαριστώ. Κυρία Φαρχάιν. Κυρία Κρόσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που βρήκατε χρόνο για να έρθετε να συζητήσουμε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε η Πέτρα Κάμερτ, γιατί ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού εμείς ε, διαπαραταξιακά συμφωνούμε σε πολλά θέματα. Τονίζω και εγώ ότι δεν είναι ιδεολογική η προσέγγιση. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι πώς οι συχνότητες που υπάρχουν περιορισμένα όμως πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η ραδιοφωνία με, από τα επίγεια συστήματα είναι το αποτελεσματικότερο μέσον για την ενημέρωση και το πολιτιστικό περιεχόμενο. Γιατί με κινητή ευρυζώνη δεν γίνεται αυτό. Ε, ε, είναι αδύνατον να, χωρίς να καταρρεύσουν τα δίκτυα να συμπεριλάβουν όλα αυτά τα, ε, τις ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Θέλουμε λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να δώσουμε προτεραιότητα σε κάποιες μεταδόσεις γιατί η δυνατότητα ε, μετάδοσης, η ικανότητα μετάδοσης είναι περιορισμένη. Και πώς ε, θα μπορέσει το ευρυζωνικό σύστημα να αντικαταστήσει τη, τα προηγούμενα, τις προηγούμενες τεχνολογίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και τις ε, ε ίνες ή άλλου ε, που θα πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο σε αυτές γιατί μακροπρόθεσμα τα, οι των δεδομένων που αναμεταδίδονται συνεχώς αυξάνονται και το καλύτερο είναι μέσα από ε, καλώδια και ίνεση άλλου. Ε, σε αυτό το τομέα λοιπόν μπορούμε να βελτιώσουμε το βασικό εφοδιασμό ούτως ώστε να ε, αυξήσουμε τη δυνατότητα μετάδοσης και μέσα από άλλα μέσα. Τονίζω και πάλι ότι δεν είναι ιδεολογικό το θέμα αλλά το πιο πρακτικό. Το δίκτυο 700 νομίζω ότι ακόμα δεν είναι στη διάθεσή μας στο βαθμό που θα ήθελαν κάποιοι. Χρησιμοποιούνται οι συχνότητες μέσα από τη ραδιοφωνία, μέσα από τη, τα κινητά μικρόφωνα. Έχουμε και άλλους τομείς χρήσης, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ε, ποια νέα ισορροπία θα υπάρχει. Υπάρχει τώρα και το δίκτυο 800 και έχουμε την Digital Dividend 1 Πολλά θα πρέπει ακόμα να δούμε, να ε, συγκεντρώσουμε εμπειρίες. Σε πολλές χώρες δεν ε, έχουν προχωρήσει τόσο πολύ και μετά θα με βάση το 800 και την εμπειρία από το Digital Dividend 1 θα μπορέσουμε να σκεφτούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Επίσης το δίκτυο δεν είναι μόνο συχνότητες 700 και 800. Πρέπει λοιπόν να δούμε ε, και άλλους τομείς ενδεχομένως ε, συχνοτήτων που μπορούν αποτελεσματικά να χρησιμοποιηθούν. Μπορούμε να υποχρεώσουμε τη, τα τηλεοπτικά προγράμματα να αξιοποιούν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τις υπάρχουσες συχνότητες. Θα αποκομίσουμε εμπειρίες και αργότερα σε εύθετο χρόνο ε, μπορούμε να σκεφτούμε το επόμενο βήμα. Χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Κρούς για την συμμετοχή σας στη σημερινή συζήτηση και διότι μας δώσατε τόσο πολλές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, πολύ σημαντικές για το μέλλον των εργασιών μας και για το μέλλον των πολιτών μας. Θα ήθελα να αφερθώ σε τρία από τα θέματα τα οποία Προστασία των ανηλίκων, ουδετερότητα του δικτύου, αξιολόγηση επιπτώσεων του ίντερνετ των πραγμάτων. Δεν θα σας ζητήσω να επαναλάβετε με περισσότερες λεπτομέρειες τα θέματα αυτά, διότι συνειδητοποιώ ότι τρεις ερωτήσεις είναι πολλές. Απλώς και μόνο, όπως ξέρετε, θα πω το εξή. Εξαρτάται αυτό από την Επιτροπή σας που πω και φέτος θα έχουμε το φόρουμ της διακυβέρνησης στα πλαίσια του ΟΗΕ για τα θέματα που μας απασχολούν και νομίζω ότι από τα τρία αυτά θέματα για το θέμα της προστασίας των ανηλίκων να έχουμε την αξιολόγηση και τα δεδομένα καθώς και τα αποτελέσματα που μπορέσαμε να επιτύχουμε τα μέτρα τα οποία εφαρμόσαμε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μας είπατε ότι γίνεται αξιολόγηση όλων των θεμάτων και αντικειμένων του ίντερνετ και πώς μπορούν να επηρεαστούν όλα αυτά μαζί με τα θέματα των ραδιοσυχνοτήτων. Αν μπορούσαμε να έχουμε όλα αυτά τα θέματα έτοιμα όταν θα συμμετάσχουμε στο φόρουμ αυτόν για την διακυβέρνηση του ίντερνετ θα ήταν πολύ χρήσιμο για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σύμφωνο με την ε, Πέτρα και τη Σαμπίνε για την πολιτική του φάσματος. Δεν θα τα επαναλάβω αυτά. Οπωσδήποτε όμως θέλω να ακούσω τις απαντήσεις και την δική σας την προσέγγιση, κυρία, αγαπητή κυρία Επίτροπε. Ε, μια... Τώρα, όταν είχαμε τους εκπροσώπους, τους εκπροσώπους της Επιτροπής εδώ, μας μίλησαν για νομική βάση και σαφείς κανόνες ε, για την ε, Ροπεάνα. Είπατε μετά ότι είναι καλό το γεγονός ότι 15 εκατομμύρια κομμάτια έχουν ψηφιοποιηθεί, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα προωθήσουμε στο μέλλον την Ευρωπαϊκή. Εσείς τι πιστεύετε. Ε, μας είπατε ότι θέλετε να ανοίξει η Ευρωπαϊκή στους πολίτες, ιδιαίτερα τους νέους ώστε να έχουν καλύτερη σύνδεση και να είναι και πιο γνωστό. Δηλαδή πώς θα γίνει, θα είναι ένα ειδικό παράθυρο, ένα window ειδικό ή πώς το βλέπετε. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Κρούς που ήρθατε. Στην εκλογική μου περιφέρεια ε, η πρόσβαση είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν είναι στο Ντάρμπισιρ ε, και γίνεται μάχη εδώ. Πώς με την ιδιωτική χρηματοδότηση για την ευρεία ζώνη. Πείθομαι δηλαδή ότι σε περιοχές όπου ε, το, η καλωδιακή δεν γίνεται, εκεί θα δοθεί προτεραιότητα στην κοινική ευρεία ζώνη. Επίσης για την εκπαίδευση ως εργαλείο όταν συζητούμε τέτοια θέματα και όταν θέλουμε να ε, αξιοποιήσουμε το ότι, είναι κάποιοι, ε, ότι ε, ο κόσμος βρίσκεται online. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες. Και μία τελευταία ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση και για τα πολλά σημαντικά θέματα που αναφέρατε. Δεν θα τα επαναλάβω. Το θέμα της ευρυζωνικό και τα θέματα που ανέφεραν οι συνάδελφοι είναι όντως πάρα πολύ σημαντικά. Θα ήθελα όμως εγώ να σας κάνω τρεις ερωτήσεις τώρα. Πρώτα απ' όλα, μία ερώτηση που θα αφορά μία οδηγία τα συγγραφικά, για τα συγγραφικά δικαιώματα που είναι τόσο σημαντικό θέμα. Μας είπατε κάτι γι' αυτό κυρία Επίτροπε και θα ήθελα να ξέρω εάν όντως σκέφτεστε κάποιους τρόπους να καταπολεμήσετε την πειρατεία στον τομέα αυτό. Γιατί πρόκειται για ε, κάτι το πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε ζωντανή τη δημιουργικότητα και τα πνευματικά δικαιώματα. Επίσης υπάρχει το θέμα της αυτοχρηματοδότησης της ε, δημιουργικής εργασίας των κυρίως σκέφτομαι τη μουσική. Σύμφωνα με αυτό το οποίο ακούμε, 30% των εσόδων στη μουσική στο ίντερνετ χάνεται εξαιτίας των πειρατών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτούς τους πειρατές του ίντερνετ. Δεν νομίζω ότι στον κυβερνοχώρο για τον οποίο μιλάμε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τη σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος. Δεύτερη ερώτηση. Το ψηφιακό χάσμα. Θα ήθελα να μου πείτε εάν στο ψηφιακό αυτό θεματολόγιο δεν θα μπορούσε να περιλάβετε προγράμματα ή πολιτών, δηλαδή υπηρεσίες ηλεκτρονικής πρόσβασης για άτομα τα οποία είναι εκτός όλων των ε, κοινωνικών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων άτομα τα οποία είναι πραγματικά αποκλεισμένα. ή πολύ νέοι, ή πολύ μεγάλοι στην ηλικία ή άτομα τα οποία ζουν στο περιθώριο της κοινωνίας θα μπορούσαν να μπορέσουν να επωφεληθούν από κάποιες τέτοιες υπηρεσίες πρόσβασης στο ίντερνετ. Επίσης, μιλήσατε για την ε, Επιτροπή Σοφών και είπατε ότι υπήρχαν τρία μεγάλα, μεγάλη διαφορετικοί άξονες του οποίους θα πρέπει να προσέξουμε στον κυβερνοχώρο. Ποιε είναι οι προτεραιότητες, σε ποιου τομεί προτεραιότητε θα μπορούσαμε ω Κοινοβούλιο να παρέμβουμε. Επίσης, για το πάρα πολύ λεπτό θέμα των τυχερών παιχνιδιών online και στην ε, ευρύτερη πρόσβαση σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αντισταθμιστεί αυτή η κατάσταση, η αυτορύθμιση ή κάτι άλλο. Έχετε σκεφτεί, έχετε προβλέψει τη θέσπιση πιο αυστηρών κανόνων για να προστατεύονται τα πιο ευάλωτα άτομα και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στους ανήλικες. Σας ξαναδίνω το λόγο κύριε Επίτροπε. Στη χαρίζω. Thank you for... Ευχαριστώ για τις ξεκάθαρες και πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρατηρήσεις, ερωτήσεις σας. Έλαβα το μήνυμά σας ότι δεν πρόκειται για ιδεολογικό θέμα εδώ και είμαι ευγνώμων που το λέτε αυτό γιατί μια τέτοια ιδεολογική αντιπαράθεση μεταξύ άλλων θα ήταν και πολύ χρονοβόρα. Πρόκειται εδώ για τη θέση της Ευρώπης, για τη, κάποια εξασφάλιση στους ε, ενεχομένους τους τομείς και σε τελευταία ανάλυση πρόκειται για τους πολίτες. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι το πρόγραμμα δεν προωθεί σαφή ε, πολιτιστικό στόχο, ούτε ε, πλήττει τους ε, οργανισμούς μεταδόσεων κλπ. Δεν έχουν αλλάξει ε, πολλά βασικά θέματα που αφορούν το γενικότερο περιβάλλον, το οποίο προωθεί τον πλουραλισμό των μέσων και την επικοινομορφία. Ε, δεν αμφισβητείται αυτό ούτε η ελευθερία των μέσων, ούτε ο πλουραλισμός. Μπορεί καμιά φορά να μην είστε απόλυτα ε, ικανοποιημένη, βλέπε ε, τα θέματα στην Ουγγαρία, αλλά ούτε εκεί ε, αμφισβητώ τον πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων. Απλώς λαμβάνω υπόψη μου τις νομικές δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν και καμιά φορά αυτό είναι δύσκολο. Κατόπιν τούτου η πρόταση απελευθέρωσης των 800 MHz είναι σόφρον, νομίζω ότι το συμφωνήσαμε. Αλλά και αναφέρομαι στην παρατήρησή σας, είναι πιο σημαντικό να ε, προωθήσουμε την κινητή ευρεία ζώνη, το διαδίκτυο, ε, πρόσβαση σε απομακρυσμένες περιοχές θα πρέπει να τους δώσουμε υψηλής ποιότητας πρόσβαση. Δεν μπορεί να υπολείπεται η Ευρώπη των άλλων περιοχών Οπότε δεν υπάρχει ως εδώ καμία παρανόηση, καμία διαφορά. Εκεί που ενδεχομένως μπορεί η πορεία μας να διαφοροποιείται είναι ότι εσείς λέτε πρώτα δώστε μας την ασφάλεια, 100% βεβαιότητα δηλαδή, και μετά θα προχωρήσουμε. Εγώ λέω από την άλλη ότι πρέπει να κινηθούμε προς τα μπρος και καμιά φορά αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να λάβουμε γρήγορα δύσκολες αποφάσεις. Και σε αυτό το φάκελο λοιπόν ο χρόνος δεν λύνει ως εκφαύματος τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και πρότεινα, κυρία Πρόεδρε, να έχουμε ε, γρήγορα την απελευθέρωση των 800 με κάποιες παρεκκλήσεις και υπογραμμίζω ότι θα έχουμε παρεκκλήσεις σε ορισμένα κράτη-μέλη που ξέρω ότι είναι αδύνατο να προχωρήσουν. Βέβαια η απόφαση μπορεί να ληφθεί. Αλλά όταν κανεί ε, ε, αν οι γείτονε ή εκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει λειτουργήσει, η λύση χρειάζεται καμιά φορά περισσότερο χρόνο. Δεν λέω δηλαδή 2013 και τέρμα τέλος, θα υπάρξουν παρεκκλήσεις με ε, στέρεα επιχειρήματα όμως. Δεν σημαίνει ότι θα πάρω με το φάσμα από ένα τομέα, αυτό που αναφέρθηκε, δεν είναι κενή η ζώνη, χρησιμοποιείται, υπάρχουν και ε, οργανισμοί ε, που χρησιμοποιούν τη συχνότητα αυτή, την ευρεία ζώνη, ε, στη δουλειά τους και το να περάσουμε από τον ένα τομέα στον άλλον, εδώ το κινητό διαδίκτυο, δεν θεωρώ ότι ε, έτσι πρέπει να γίνει. Θα εξισορροπήσουμε τις μελλοντικέ ανάγκες, αυτό περιμένετε και από μένα. Να λάβω υπόψη μας πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στο μέλλον και θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει. Εδώ εσείς ζητάτε σαφήνεια για να μην διαιωνίζουμε μια κατάσταση και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να εξισορροπήσουμε τις μελλοντικέ μας ανάγκες λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία του διαδικτύου. Το διαδίκτυο πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και συνδέεται και με τις προσδοκίες των πολιτών. Η σημασία του διαδικτύου λοιπόν δεν αμφισβητείται. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να προβλέψουμε πολιτιστική προστασία και να προωθήσουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό στον κόσμο. Σε ό,τι με αφορά πρέπει να παρακολουθήσουμε πώς χρησιμοποιείται το φάσμα ώστε να ξέρουμε ότι ε, αποτελεσματικά χρησιμοποιείται. Και ο χρήστης ο μελλοντικός και ο χρήστης, ο οποίος μπορεί να απειλείται, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με τρόπο αποτελεσματικό. Και αν δεν γινόταν αυτό στο παρελθόν, τώρα είναι αδύρυτη ανάγκη. Και εξεπλάγει πραγματικά, ακούγοντας όλες αυτές τις προσδοκίες για την ενδυνάμει χρήση αυτού του διαδικτύου, τη διακυβεύεται, θα αρχίσουμε με ένα τσουνάμι. Δεν είναι λοιπόν θέμα καλής προαίρεσης. Μέσα σε, εξι... σε τρεις μήνες ε, όμως ε, είναι αδύνατο να εξηγήσουμε όλες τις λεπτομέρειες της νέας πραγματικότητας. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε θα κινηθούμε προσεκτικά. Εγώ ζητώ όλου, από όλους να γνωρίζουν ότι θα κρυθούν με βάση την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους και έτσι θα κινηθούμε προς μια λύση που θα προβλέπει και παρεκκλήσεις εξαιρέσεις που όμως θα στηρίζονται όπως σας είπα σε πολύ ε, σαφή και έγκυρα επιχειρήματα ιδιαίτερα όταν πρόκειται για χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με γειτονικέ χώρες και πραγματιστική προσέγγιση, παρέκκληση μόνο εμπεριστατωμένη και λογική. Προσπερνώ κάποια θέματα ε, είπαμε για την ουδετερότητα του δικτύου. Νομίζω ότι και πέρσι ήταν ε, σαφής η παρέμβασή μου. Θα μπορούμε να ε, δικαιολογούμε περαιτέρω ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν θα... Ε, αν δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, δεν είμαι υπέρ των κανονιστικών, ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Και βέβαια υπάρχει και θέμα με τους ανταγωνιστές. Ε, τους, τους εταιρείες. Ε, αν εξετάσουμε ε, όλα αυτά τα θέματα, τότε συμφωνώ. Ακόμα δεν έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειαζόμαστε αλλά νομίζω ότι αν λάβουμε δράση θα πρέπει να κινηθούμε με διαφάνεια ποιότητα υπηρεσιών για να βοηθήσουμε τους πελάτες, να έχουμε υποχρεώσεις ε, μη διακριτικές για τους παρόχους του διαδικτύου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και πρέπει να σας το πω, γιατί κάποιος μίλησε για μεγάλες επενδύσεις που χρειάζονται για την εξάπλωση της ευρεία ζώνης. Το συζητήσαμε, συζητήσαμε για 200-300 δις ευρώ. Όχι αύριο, αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν είναι ψηλολόγια και όλοι περιμένουν να υπάρξει συμφωνία. Υπάρχουν όμως κάποιοι σε αυτή που ενδιαφέρονται για αυτή τη διαδικασία Αλλά ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι αν δεν αναλάβουμε δράση θα ε, χάσουμε ε, ως Ευρώπη τη θέση μας παγκοσμίω. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε ό,τι χρειάζεται για τις επιγραμμικές τεχνολογίες και διαδικασίες. Οι περιεχομένου είναι δραστήριοι στη Silicon Valley και αν δεν αναλάβουμε δράση τώρα, ε, ε, θα αγοράζομαι μόνο από τις δύο πλευρές ε, χωρίς να αξιοποιούμε αυτά από τις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται και στη, στο επίπεδο της οικονομίας. Κάλεσα λοιπόν τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιριών τηλεπικοινωνιών κάποιοι που ασχολούνταν. Αυτή ήταν μια ομάδα, η άλλη είναι η πάροχη περιεχομένου, μια άλλη ομάδα είναι η ε, ραδιοφωνικοί οργανισμοί και οι κατασκευαστές τέλους. Τέσσερις ομάδες. Είπαμε να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι σε ανώτερο ε, επίπεδο και ο Steve Jones ε, συμμετείχε και τους είπα ότι από εσάς εξαρτάται, ε, θεωρώ ότι δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων, εσείς που έχετε τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, ενέχεστε σε όλες αυτές τις εξελίξεις, οπότε θα πρέπει να συζητήσετε με τους αρμόδιους τι διακυβεύεται στον τομέα σας. Να είστε δημιουργικοί πέρα από στερεότυπα, νέα επιχειρηματικά μοντέλα δεν, τα παλιά δεν αποτελούν λύση πολλές φορές. Άρα λοιπόν ας καθίσουμε όλοι μαζί, ας δουλέψουμε σε ομάδες εσείς. Θα δείτε το διακύβευμα κάθε φορά. Και θα δημιουργηθούν έτσι νέα ε, δημιουργικά επιχειρηματικά μοντέλα, τα οποία και στις 13 Ιουλίου ε, σε μια νέα συνεδρίαση θα δούμε αν όλα αυτά ε, είναι λειτουργικά. Τι διακυβεύεται. Σωστά το είπατε, δεν μιλάμε μόνο για καλωδιακή, για ίνες ή άλλου, ή χαλκού, ή δορυφόρους ή οτιδήποτε άλλο. Πρόκειται για μια ποικιλομορφία και όλοι συμμετέχουν. Είναι ένα μείγμα και δεν μπορεί να λειτουργήσει αν κάποιος μόνο ε, πληρώνει το λογαριασμό. Μάλιστα πιεζόμεθα από το χρόνο. Και πάντα εξηγώ ότι σε τελευταία ανάλυση όταν μιλάμε για την οικονομία και τη στρατηγική της Ευρώπης 2020, ε, αυτός είναι ένας έξυπνος τρόπος για να ε, λύσουμε αυτό το κομμάτι της οικονομικής μεγέθυνσης, καταπολέμησης της ανεργίας κλπ. Ε, περιμένετε λοιπόν μέχρι τις 13 Ιουλίου και οπωσδήποτε θα επανέλθω για να σας ενημερώσω. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αν δεν έχουμε επιτυχία θα πρέπει εγώ να αναλάβω δράση, αλλά αυτή είναι η ίστατη λύση. Δεν φοβάμαι να αναλάβω δράση, αλλά καλύτερα θα ήταν να λειτουργήσουν οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι με τις καινοτόμες, τις δημιουργικές τους προσεγγίσεις. Τώρα για την πειρατεία και τα διανοητικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία και, και την Ευρωπαϊκή. Διστάζω λίγο να μιλήσω για μεγάλη επιτυχία μέχρι τώρα. Βέβαια, ότι πλασιάστηκαν, ότι έχουμε 15 εκατομμύρια κομμάτια είναι καλά, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα. Ε, ε, ότι δεν, δεν, δρά ακόμα υποστηρικτικά ε, ο Ευρωπαίανα. Δεν έχω μιλήσει όλα τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν μπορώ ε, να τα εξηγήσω όλα αυτά στους πολίτες. Βέβαια, ο περασμένος ε, αιώνας ήταν διαφορετικός και έδωσε πάρα πολλές καταπληκτικές καινοτομίες ε, τώρα πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τα καινούργια και δεν μιλάω μόνο για την πειρατεία βεβαίω και είναι ανεπίτρεπτη και παράνομη και πρέπει να καταπολεμηθεί η πειρατεία αλλά αν δεν, λύσουμε, αν δεν πιάσουμε στη ρίζα το πρόβλημα και λύσουμε μόνο το σύμπτωμα και καταπιαστούμε με το σύμπτωμα αυτό δεν είναι σωστό θα πρέπει λοιπόν να λυθεί το πρόβλημα ε, αποτελεσματικά. Κλείσει δηλαδή αυτή η στρόφιγγα. Αυτό είναι υποχρεωτικό, πρέπει να προχωρήσουμε ε, σε αυτό το δρόμο και αυτό που είναι σαγηνευτικό στην τεχνολογία είναι ότι εντωμεταξύ υπάρχουν και ομάδες καλλιτεχνών, ε, συγγραφέων που χειρίζονται με τον τρόπο τους τις νέες πληροφορίες και αξιοποιούν τις νέες ευκαιρίες και μετά ε, έχουν κάνει ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό θα πρέπει να ανταμείβονται και θα πρέπει αυτό να γίνεται άμεσα, όχι στο απότερο μέλλον. Και δεν μιλάμε για τα μεγάλα αστέρια, μιλάμε για τους ανθρώπους που κάνουν την πρωτοπόρα δουλειά, την οποία όλοι εκτιμούμε και θέλουμε να συνεχιστεί η νομική βάση της Ευρωπαϊάνα και τι παίζεται, τι διακυβεύεται τώρα. Πρέπει να έχουμε μια στέρεη βάση για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊάνα, γιατί δεν μιλάμε μόνο εδώ για τη νομική βάση, μιλάμε για τον τρόπο της χρηματοδότησης και όχι μόνο για τα επόμενα δύο χρόνια ας πούμε. Πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και θα πρέπει να προωθήσουμε την Ευρωπαϊκή με πολύ πιο στοχευμένο τρόπο, λαμβάνοντα υπόψη τα όσα διακυβεύονται τώρα. Τώρα, η βελτίωση της ευρυζώνης, ε, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός ε, είναι ε, πολύ σημαντικό, είναι μια προτεραιότητα δηλαδή που συμπεριλαμβάνεται Γνωρίζω ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε περισσότερο για να ενημερώσουμε για την Ευρωπαϊκή, να την κάνουμε πιο ελκυστική, να είναι πιο ελκυστικό το πρόσωπό της από ό,τι μέχρι τώρα. Ε, έχουμε ε, επιτροπές ε, εκτός από την Επιτροπή των Σοφών και η δεύτερη επιτροπή έκανε εξαιρετική δουλειά και είμαι ευγνώμων. το πρώτο βήμα είναι Α, και επίσης είμαι και πολύ ευγνώμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που επικούρησε την Κομισιόν και από κοινού ε, αποφασίζομαι τα βασικά και μετά τα βελτιώνουμε ακόμη περισσότερο. Ε, εκαλυφθήκατε όλοι από τις απαντήσεις. Εσείς, παρακαλώ, Τσέλγκα. Όλοι ξέρουμε πόσο μεγάλα είναι τα προβλήματα και επίσης ότι δεν είναι εύκολο να ευρεθεί για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή η κατάλληλη λύση. Τι ερώτησα εγώ. Μετά από διάφορες συναντήσεις τους ε, η Επιτροπή των Σοφών ζήτησε νομική βάση παγιωμένη. Υπάρχει απάντηση. Πώς προσπαθείτε ε, να το λύσετε. Ξέρουμε ότι είναι σημαντικό να λυθεί. Το ερώτημα είναι τι κάνετε. Τι ιδέες υπάρχουν. I'm pushing my colleague. Ε, Σπρώχνω τους συναδέλφους και ελπίζω ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση στα πλαίσια της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και ελπίζω ότι σύντομα, σύντομα στο μέλλον θα έχουμε ένα μέσον ευέλικτο και σίγουρο. Το επόμενο βήμα λοιπόν θα είναι αύριο να το έχουμε στη μήνυση δέξη των πιο ενδιαφέροντων θεμάτων για να το λύσουμε. Πολύ ωραία. Ελπίζουμε όταν σας ξαναδούμε να έχει λυθεί το πρόβλημα. Να είστε λοιπόν ανυπόμονοι, όπως και εμείς, για να προχωρήσουν τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπη. Ξέρω ότι είστε βιαστικοί, σας ευχαριστούμε και καλή τύχη. So. Σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη. Μία ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Ό,τι είναι σημαντικό στην προοπτική του 2020 η συμβολή της Ευρώπης για την απασχόληση η συντάκτρια, θα, κυρία Νεβεντάλοβα, θα μας παρουσιάσει την εργασία της μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να πω ότι η νέα γενιά σήμερα είναι πιο καλά εκπαιδευμένη, ε, πιο μορφωμένη, αλλά έχει πολύ άσχημη ε, δυνατότητα απασχόλησης. Οι νέοι διαρωτώνται σήμερα αν έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να βρουν μια θέση εργασίας. Αγγλικά μιλάει η γυναίκα. Αγγλικά μιλάει. Α, ε, στην αρχή μίλησε Σλοβάκικα, γι' αυτό τρελάθηκα. Ε, ε τώρα... Λοιπόν, θα Πρέπει να συνδέσουμε την σωστή κατάρτιση με την εργασία και την απασχόληση. Η... Τα αρμόδια υπουργεία πρέπει να συνεργαστούν σωστά σε κάθε χώρα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορούν επακριβώς να πούν τι δεξιότητες στο μέλλον θα καταστούν απαραίτητες. Παράλληλα, είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι ο πληθυσμός, ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γυράσκει και γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν εξειδικευμένες δεξιότητες και σε αυτό το τομέα. Οι σημαντικότερες δεξιότητες που πάντα θα είναι αναγκαίες είναι οι τεχνολογίες ε, της πληροφορίας. Όσοι είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό το τομέα, ε, πιο εύκολα θα βρίσκουν απασχόληση. Οι γλώσσες είναι σημαντικές επίσης. Σήμερα κάποιος λένε ότι πρέπει να ξέρει όχι μία αλλά δύο και τρεις ξένες γλώσσες. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, το θέμα των γλωσσών των μεταναστών. Καλό είναι να υποστηριχθεί η διδασκαλία και αυτών των γλωσσών ή και σε αυτές τις γλώσσες, διότι αυτό εμπλουτίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι πράσινες δεξιότητες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, στην οικολογία και επίσης συνδεδεμένα με όλα αυτά είναι και η δημιουργία των πράσινων θέσεων εργασίας. Όπως είπε η συνάδελφος Άξελα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη μας και εκείνες τις δεξιότητες που ε, είναι γενείς στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στον τομέα της βιοτεχνίας, των υπηρεσιών που εξαφανίζονται. Ε, είναι απαραίτητο να υποστηριχθούν και αυτές. Προσωπικά είμαι πεπισμένη ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την επίσημη και άτυπη εκπαίδευση ε, και ε, μέσα από σεμινάρια, διασκέψεις επίσης αποκτώνται δεξιότητες που ίσως με άλλο τρόπο δεν μπορούν να αποκτηθούν. Επικοινωνιακές ικανότητες ε, η ικανότητα έκφρασης ε, και όλα αυτά. Επίσης ε, θέλω να αναφερθώ στην υποστήριξη της διαβίου μάθησης. Επίσης υποστηρίζω τη γενική αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση. Όλα αυτά είναι τομείς που επηρεάζουν πάρα πολύ την αύξηση της απασχόλησης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για νέους ανθρώπους. Επίσης, να προσπαθήσουμε στον τομέα της αναγνώρισης της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι η μέση εκπαίδευση δεν την χάνει τόσο μεγάλης κοινωνικής αποδοχής όσο το πανεπιστημιακό πτυχίο. Και οι δύο βαθμίδες όμως είναι πολύ σημαντικές και επίσης η ισότητα ανδρών γυναικών είναι σημαντική σε όλες τις δεξιότητες και σε όλους τους τομείς θα πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη γιατί Πρέπει παντού να φροντίσουμε για την ισότητα των δύο φύλων. Επίσης, ε, ένταξη ανθρώπων με αναπηρίες σωματικές ή ψυχικές. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η γνωμοδότησή μας έχει ολοκληρωθεί ήδη και ελπίζω ότι σύντομα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Εγώ ε, ευχαρίστως να συναντήσω και να συζητήσω τους σκιώδεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα ε, χρειαστεί να παρέμβει η Κομισιόν ή μήπως το επιθυμεί. Θέλετε να πείτε κάτι τώρα, Κομισιόν. Όχι, όχι πολύ, λιγάκι, σύντομα. Την επόμενη φορά, την επόμενη φορά να έχει ετοιμαστεί και τότε θα μας τα πει όλα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Παδία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κατερίνα Νεβεντέλοβα για αυτή την ε, σύντομη, πολύ συγκεκριμένη παρέμβασή της για τις νέες δεξιότητες και τις θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι για κάποιες ε, έννοιες θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Η τερολογία είναι σημαντική. Μας είπε για το ποιες θα είναι οι νέες δεξιότητες και τα νέα προσόντα τα επαγγελματικά. Πριν από αυτό θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει πρώτα να ξέρουμε ποιε θα είναι οι νέε θέσει επασχόλησης που θα δημιουργηθούν. Πριν να ξέρουμε λοιπόν πώ θα καταρτήσουμε του ανθρώπου, του νέου κυρίω, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις νέες θέσεις επασχόλησης. Διότι μιλάμε για πράσινες θέσεις εργασίας, λευκές θέσεις εργασίας για τους μεγαλύτερους και θα πρέπει να αποσαφινιστούν αυτές οι έννοιες. Πιστεύω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει το θέμα αυτό να το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Επίσης, έκανα ένα σχόλιο για την παιδεία, για την εκπαίδευση, την επίσημη, επίσημη και ούτως ή άλλως θα πρέπει να πούμε το εξής όποια και να είναι η θέση επασχόληση, Όποιε και θα είναι οι νέε δεξιότητε που θα δημιουργηθούν, ό,τι έχει σχέση με την καινοτομία και την δημιουργικότητα και με την, ε, το επιχειρήν θα πρέπει να τα τονίσουμε εδώ γιατί είναι πολύ σημαντικά. Και όταν δούμε ποιε θα είναι αυτέ οι νέε θέσει απασχόληση και οι δεξιότητε για να μπορέσουμε να τι επεξεργαστούμε περαιτέρω, θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το θέμα τη κατάρτιση των εκπαιδευτών. Ευχαριστώ. Έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Μίχαλ Ντόιτς από την Κομισιόν θέλει κάτι να πει. Ε, ε, ε Γιατί σας βλέπω απογοητευμένο. Έχετε έτσι μια, ένα ύφος απογοητευμένο. Αν θέλετε να λάβετε το λόγο, ευχαρίστως. Εγώ για σας το είπα, μήπως δεν ε, θέλατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι ο κύριος Τέτσο από την Άκτα, αλλά είμαι εκπρόσωπος της, Επιτροπής, της ε, Διεύθυνσης Απασχόλησης και για πρώτη φορά έρχομαι εδώ. Μην πει, δεν ε, σκέφτηκα σε αυτό το στάδιο να λάβω το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής. Ελπίζω όμως ότι σε μία επόμενη συνεδρίασή σας θα συζητηθεί έκθεση με μεγάλη ευχαριστή εγώ και συνάδελφοι της Γενικής Διευθυνσής μου θα λάβουμε το λόγο. Επειδή ήταν πρώτη φορά που είστε εδώ, γι' αυτό είπα αυτά που είπα. Πολύ καλά. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Ο κύριος Βάτιμο. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση της Κατερίνας μου φαίνεται ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα για το θέμα αυτό των νέων απασχολήσεων. Δεν θα πρέπει να επικεντρωθούμε μόνο στην πληροφορική και στις γλώσσες. Ναι, είναι δύο σημαντικά θέματα αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και νέοι πτυχιούχοι ε, της φιλοσοφικής που δεν βρίσκουν δουλειά. Έρχονται σε μένα και τους λέω μάθετε ξένες γλώσσες και μάθετε χρησιμοποιείτε το κομπιούτερ. Αλλά στην κοινωνία μας υπάρχουν, ε, υπάρχει ανάγκη να αναπτύχουν και δεξιότητες βιοτεχνίας αν θέλετε δεν ξέρω αν ε, υπερβάλλω, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι στη μέση εκπαίδευση τέτοιου είδους ε, θέματα δεν διδάσκονται. Δηλαδή, κάποια πολύ απλά αντικείμενα δεν ξέρει κανείς τα χειρίζεται και μόλις πάθουν την παραμικρή βλάβη τα πετάει στα σκουπίδια. Σήμερα ξέρουμε ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι ε, καλλιεργούν λαχανικά στους ταράτσες τους, στα μπαλκόνια τους, για να έχουν τα δικά τους λαχανικά. Άρα υπάρχουν δυνατότητες να επανέλθει κανείς στην ε, γεωργία. Δηλαδή να προσπαθήσει κανείς ε, στο σημερινό μας υλικό κόσμο να είναι πιο προτεκτικός, να μην ακολουθεί πάντα το ότι αγοράζω, χαλάει, το πετάω, τελείωσε. Δεν λέω ότι ο καθένα θα πρέπει να μάθει μια τέχνη, αλλά για να ράψει κανεί ένα κουμπί μεταξύ των νέων σήμερα είναι όλο και πιο δύσκολο. Επίση, όλο και λιγότερε μοδίστρε υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν και κάποια επαγγέλματα τα οποία τα αποφεύγουμε σήμερα. Να μην το ξεχνούμε αυτό, διότι όλοι αντιμετωπίζουμε από την έλλειψή του τέτοιου είδου καταστάσει. Ο κύριος Τσβέερ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Υποθέτω ότι ποτέ τα σχολεία δεν ήταν σε τόσο δύσκολη θέση όπως σήμερα. Διότι έχουμε διαφορετικών ειδών οικονομίες, προβιομηχανική, βιομηχανική, κλασική, μεταβιομηχανική, Τη κοινωνία της πληροφορικής, μεταπληροφορική. Δύσκολα λοιπόν μπορεί και το σχολείο να βρει τι ε, επόμενε μελλοντικέ ανάγκε ε, για νέε δεξιότητε και θέσει εργασία. Και θα πρέπει πάντα να υπάρχει μια σύνταξη παιδεία και εργασία. Ο κόσμο εργασία δεν θα πρέπει να είναι μέσα από το σχολείο και τούμπαλιν. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει το σχολείο να δει τι χρειάζεται η μελλοντική κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ νομίζω ότι στην πρόταση πρέπει να αναφέρομαι ότι πρέπει και η επιχειρηματικότητα, για παράδειγμα, να διδάσκεται στο σχολείο. Οι νέοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν δράση οι ίδιοι, να κάνουν κάτι. Έχω δει ανθρώπους που έχουν αναλάβει να ανοίξουν ένα μικρό κατάστημα. Μικρό μεν, λειτουργικό όμως αυτές οι δυνατότητες, τα ταλέντα που έχει ο καθένας πρέπει να βγαίνουν στην επιφάνεια και να αξιοποιούνται. Και από νωρί θα πρέπει και να δίνουμε στους νέους ε, αυτές τις δυνατότητες. Να μην αναλαμβάνουν εκείνοι, να γίνονται ε, επιχειρηματίες. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα στο σχολείο, αλλά πολλά μπορούν να προσφέρουν εδώ. Γι' αυτό χρειάζονται και οι καθηγητές που θα προσεγγίζουν με αυτόν τον τρόπο τα θέματα και θα μαθαίνουν τα καινούργια αυτά στοιχεία τα παιδιά αυτό. Στη... Στο μέλλον θα μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε εδώ αυτό το θέμα της κυρίας Νεβεντάλοβα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ Κατερίνα και σου εύχομαι επιτυχία στην έκθεση. Προχωρούμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ο συνάδε... η συνάδελφος Κώστα ε, είναι η συντάκτερη της γνωμοδότης να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως θα γνωρίζετε, όλοι είναι συντάκτες γνωμοδότης, ξέρετε ότι η γνωμοδότηση δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 1500 ε, χαρακτήρες στο κομπιούτερ. Η έκθεσή μου λοιπόν είναι πάρα πολύ συνοπτική, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ε, θέματα για τα οποία ήδη έχω αναγγείλει κάποιες τροπολογίες. Δεύτερον, είμαι ανοιχτή σε οποιαδήποτε υπόδειξη εκ μέρους σας. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω στην έκθεση αυτή είναι η πάρα πολύ στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ επένδυσης σε θέματα πολιτιστικά και παιδείας, καταπολέμησης της στόχες και του κοινωνισμού αποκλεισμού και ανάπτυξη μια κοινωνία. Κατά την άποψή μου, αυτό το θέμα δεν έχει αναλυθεί πάρα πολύ σωστά στην έκθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είναι από τα σημεία κίνηση τη δική μου έκθεση. Και θα ήθελα να ζητήσω στα εθνικά σχέδια μεταρρύθμιση τα κράτη-μέλη να αναγγείλουν επενδύσει σε αυτό το νομέα που επαναλαμβάνω πολύ σημαντικέ για την ανάπτυξη. Δεύτερη παρατήρηση. Θα ήθελα να συστήσω στα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν την εγκατάλειψη του σχολικού συστήματος σε πολύ πρώιμο στάθμο, διότι αυτό οδηγεί στον κοινωνικό αποκλεισμό. Θα πρέπει να προβλεφθούν λοιπόν ε, συστήματα στα οποία να συμπεριλαμβάνονται όλες οι ομάδες του πληθυσμού, ε, μαθητεία, ειδικά μαθήματα για αναπήρους κτλ. Τρίτον, είναι απαραίτητο να υπάρχουν μόνιμα και διαρκή προγράμματα κατάρτισης και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους στα πλαίσια του προγράμματος που προβλέπεται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων για να μπορέσει κανεί να επιτύχει μια καλή θέση εργασίας. Στα νηπιαγωγεία νομίζω ότι για το 2020 θα πρέπει να μπορούν να γίνονται σχεδόν όλα τα παιδάκια αποδεκτά δεκτά συγγνώμη, από τα τέσσερα τους. Επίσης, ήδη από τότε να προβλέπονται αθλητικές ε, δραστηριότητες, γλώσσες και οτιδήποτε μπορεί να τα βοηθήσει. Τα θέματα τα πολιτιστικά και τα θέματα της δημιουργικότητας, τα προγράμματα ε, ε, κοινωνικής ε, συμπερίληψης όλων των ομάδων, ακόμη και των πιο ευάλωτων στην κοινωνία, είναι σημαντικά. Ακόμη και μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων θα πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση, διότι δεν είναι εύκολο να έχει κανείς ε, πρόσβαση στα προγράμματα Far Youth on the Move. για θέματα παιδείας ή απασχόλησης. Επίσης θα ήθελα να πω πόσο σημαντικά είναι τα προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για ανήλικου ή ενήλικους σε συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τη συνδρομή κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταμεία. Επίσης θα πρέπει όλες οι γνώσεις και τα προσόντα ατόμων που είναι σε ένδια να μπορέσουν να αξιολογηθούν Πάντα θεωρούμε ότι είναι δικαιούχοι κάποιων προγραμμάτων, αλλά πάντα πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι, οργανώσει που έχουν πολύ καλά προσόντα ή δεξιότητε, ακόμη και για να διδαχθούν κάποια επαγγέλματα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένω. Επίση, ο εθελοντισμό θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να μπορέσουν να μειωθούν τα ποσοστά φτώχεια. Πρόκειται για θέματα τα οποία ανέφερα πάρα πολύ ε, συνοπτικά. Σας είπα ότι ήδη κατέθεσα τροπολογίες για την κατάρτιση των εργαζομένων, για καλύτερη συμπερίληψη όλων στην κοινωνία που θα πρέπει να έχει καλύτερη κατάρτιση, καλύτερη εκπαίδευση. Υπάρχει το θέμα των ε, επίσημων ή άτυπων δραστηριοτήτων και θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις όσων αυτών των αλλαγών στη φτώχεια. Διότι από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχουν συγκρίσιμες στατιστικές ε, μεταξύ των κρατών μελών για το πόσο αποτελεσματικές είναι οι δράσεις, κυρίως, κυρίως για να μπορέσει κανείς να ξεφύγει από την φτώχεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ανίβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Κώστα. Θα ήθελα να τονίσω μερικά πράγματα. Πρώτον, το θέμα της πρώιμης εγκατάλειψης του σχολείου. Όταν έγραφα την έκθεση για την προσχολική ηλικία, είχα δει ότι είναι σημαντικό να αποφύγουμε το φαινόμενο της πρώιμης εγκατάλειψης των σχολείων. Γι' αυτό νομίζω θα έπρεπε να το αναφέρουμε και αυτό θα ήταν παράληψη. Γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά κάτι άλλο που το ανέφερε μεν η κυρία Κώστα αλλά πρέπει να το τονίσουμε αλλιώς είναι το όλο θέμα της μετανάστευσης. Αυτοί που ξεφεύγουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανέχεια και που στη Βρετανία τις λέμε εθνοτικές μειονότητες είναι βασικά μετανάστες αυτό πρέπει να τονιστεί γιατί εκείνοι είναι αυτοί που αποκλείονται κοινωνικά. Μπορούμε να ζητήσουμε ειδικά μέτρα παιδείας για αυτούς όπως κάποια εκπαίδευση στη γλώσσα τους, να έχουν κάποιες περισσότερες ευκαιρίες μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τόσο περιθωριακή όσο είναι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε ναι, φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αν και συνδεδεμένες. Είναι εδώ κάποιος από την Επιτροπή Απασχόλησης, ο κύριος Χάλτους. Εδώ είναι? Όχι, δεν είναι. Ωραία. Κύριε Αντεκώστα. Εντάξει, το κλείνουμε λοιπόν το θέμα εδώ και εσείς θα ανασκουμποθείτε για την έκθεση. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε πολύ. Πού είναι η Χάνου Τακούλα. Δεν είναι εδώ. Ο, Χάνου. το, είναι στο Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Μπορεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορεί να αναλάβει άλλος. Θα συζητήσουμε ή όχι για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και ας μείνει ο κύριος Τάκουλα εδώ. Έχει κανείς να πει κάτι πριν μιλήσει για το θέμα κύριο Στάκουλα. Όχι. Πρέπει, είναι παράδοξο ακούγεται αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν καταλαβαίνει κανείς εύκολα τι εννοεί, αλλά είναι στο στόμα όλων και πρέπει να εξοικειωθούμε. Α, ο κύριος Κέλλη θα μας μιλήσει για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό, όπως είπατε κι εσείς, για να αντιμετωπίσουμε την τωρινή κατάσταση, να διασφαλίσουμε ότι αντλήσαμε τα διδάγματα που έπρεπε. Και οι χώρες θα πρέπει να εξετάσουν τις πολιτικές τους και τους προϋπολογισμούς τους. Αυτό είναι ζωτική σημασία. Εγώ για τη χώρα μου μπορώ να πω ότι αν είχαμε τα τελευταία χρόνια ε, αξιοποιήσει την ιδέα του ευρωπαϊκού εξάμεινου, τότε πολλές διασπαθήσεις θα είχαν αποφευχθεί και κάποιοι εμπειρογνώμονες εκτός της χώρας μου θα έλεγαν προσέξτε εδώ για να αποφευθεί κάποια καταστροφή. Έτσι λοιπόν είναι μέτρα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα διασφαλίσουν ότι στο τέλος της ε, κρίσης δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα ε, διασπάθησης κονδυλίων. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ κυρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί ήρθα με τέτοια καθυστέρηση. Υπάρχουν σημαντικά θέματα που συζητιούνται στο Κοινοβούλιο, και είναι και αυτό σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Συνεργασία είναι για τη δική μας Επιτροπή κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, το γνωρίζουμε αυτό, γιατί δυστυχώς πολύ συχνά η Κομισιόν θεωρεί ότι η εκπαίδευση είναι κάτι το προφανές, τόσο προφανές που ούτε το αναφέρει στις εκθέσεις της. Αν όμως θέλουμε μία, ένα εργατικό δυναμικό ποιότητας, είναι τελείως απαραίτητο να υπάρχει πανενοσιακή ποιοτική εκπαίδευση παιδεία και γι' αυτό χρειάζεται ακριβώς αυτή η ποιοτική μάθηση. Άρα πρέπει γενικά η παιδεία από, από την μικρότερη δυνατή ηλικία να καταλάβουμε ότι πρέπει να τύχει επένδυσης να είμαστε σε θέση δηλαδή να παραγάγουμε μια ένα ποιοτικό εργατικό δυναμικό. Η σημασία λοιπόν της παιδείας και της εκπαίδευσης μεταξύ άλλων και των διδασκάλων είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα. Αν δεν έχουμε καλούς δασκάλους δεν μπορούμε να έχουμε καλούς μαθητές. Με άλλα λόγια θα έπρεπε να δηλώσουμε στεναρά προς την Κομισιόν ότι Κυρίες και κύριοι της Επιτροπής, αν θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη μην ξεχνάτε την παιδεία και την εκπαίδευση γιατί είναι το κλειδί, το κλειδί για την βιώσιμη ανάπτυξη. Ποιότητα και διαβίου μάθηση είναι τα κλειδιά. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σημαντικό σε αυτήν τη φάση, βλέποντας το μέλλον, να γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Υπήρχαν και χειρότερες εποχές από αυτήν την κρίση, παραδείγματο χάρη αμέσω μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, πολλές χώρες μέλη, τωρινές χώρες μέλη, είχαν τότε σημαντικά χρέη που έπρεπε να πληρώσουν μετά τον πόλεμο, οι υποδομές ήταν κατεστραμμένες και η αύξηση του ΑΕΠ ήταν στο μηδέν. Οι προπάτορες της Ευρώπης κατάλαβαν, είχαν καταλάβει ότι η εκπαίδευση και η παιδεία θα είναι το κλειδί τα επόμενα 20-30 χρόνια. Αλλά και στην τωρινή κρίση υπάρχει υπερχρέωση και πρέπει και πάλι να κάνουμε επενδύσεις στην παιδεία διότι η παιδεία και η εκπαίδευση θα φέρουν καρπούς για να αν θέλουμε η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική διεθνώς. Κυρία Πρόεδρε, δύο λόγια ακόμη για τη στρατηγική 2020. Δυστυχώς δεν λέμε πολλά για την παιδεία και την εκπαίδευση. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα αυτό, μεγαλύτερη προτεραιότητα. Πιο φιλόδοξους στόχους, ας πούμε. Να μειωθεί ο αριθμός όσων εγκαταλείπουν νωρί το σχολείο στο 10% μόνο. Αν και ο αριθμός αυτός είναι και αυτός υψηλός. Δεν νομίζω ότι πρέπει ούτε ένας μαθητής να εγκαταλείπει το σχολείο. Δεν συνάντησα βέβαια ούτε έναν Υπουργό Παιδείας στην Ευρώπη που να μου δηλώσει ότι υπάρχουν πάνω από 10% μαθητών που εγκαταλείπουν νωρί το σχολείο. Λένε ότι όλοι έχουν ήδη πετύχει το στόχο του κάτω του 10% εγκατάλειψης αν έχουμε επιτύχει αυτόν τον στόχο τι τον θέτουμε θα μας λένε αλλά εγώ δεν το πιστεύω Νομίζω ότι εφαρμόζονται διαφορετικά πράγματα σε διαφορετικές χώρες και εγώ ξέρω από την δική μου χώρα τη Φιλανδία ότι αυτό που συζητιέται είναι ότι κάθε μέρα πέντε μαθητές και φοιτητές αποκλείονται από την παιδεία. Άρα το κόστος που, με το οποίο θα επιβαρύνουν την κοινωνία είναι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Αν θα μπορούσαμε έναν έστω να απασχολήσουμε θα λυνόταν το πρόβλημα. Σε αιτήσιο δε επίπεδο στην κοινωνία της Φιλανδίας ο αποκλεισμός των νέων κοστίζει 2 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο είπαμε και άρα ακόμη και ένας που εγκαταλείπει το σύστημα είναι κάτι το ιδιαίτερα βαρύ. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτούς τους ανθρώπους να βρουν τη θέση τους στην κοινωνία. Γιατί δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα μετράμε μόνο με οικονομικά μέτρα αλλά και με πνευματικά και με διανοητικά. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να οικοδομήσει την Ευρώπη. Η βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό είναι το μήνυμά μας προς την Κομισιόν, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και ως προς την παιδεία. Επομένως, παρακαλώ, βάλτε περισσότερο την παιδεία στα προγράμματά σας. Γιατί είναι κάτι που θα φέρει καρπούς. Κυρία Πρόεδρε, πάνω κάτω αυτές είναι οι σκέψεις που ήθελα να εκφράσω και που γράφω εδώ στο εγγραφό μου και θα συνεχίσω τη συζήτηση όποτε και όπως θέλετε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, είμαι ο σκιώδης συζητητής για το ζήτημα αυτό, για το EPP. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Τάκουλα, για όλα όσα είπε και να προσθέσω και εγώ μερικά σημεία στην πρώτη συζήτησή μας σε σχέση με το τι, διακυβε... διακυβεύεται στην ε, τοποθέτηση αυτής της Επιτροπής μας και πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που μας δίνεται. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας σε σχέση με τους υψηλούς στόχους που πρέπει να έχουμε στα θέματα της παιδείας να υπενθυμίσω ότι εξίσου υψηλούς στόχους είχαμε και την προηγούμενη δεκαετία με την στρατηγική της Λισαβόνας. Και οι στόχοι αυτοί δεν επετεύχθησαν. Και όταν καταστρώσαμε τη νέα στρατηγική μας για το 2020, αρκεστήκαμε να πούμε ότι δεν πετύχαμε τα προηγούμενα, πάμε τώρα να πετύχουμε κάποια περισσότερα. Το γεγονός ότι πλέον καθιερώνεται αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο για το συντονισμό των πολιτικών μας δίνει την ευκαιρία να παρακολουθούμε την πρόοδο σε σχέση με τους στόχους που έχουμε θέσει και βεβαίως να είμαστε ιδιαιτέρως επικριτικοί αν κρίνουμε ότι, και έγκαιρα αν κρίνουμε ότι οι στόχοι αυτοί δεν βλέπουμε να επιτυγχάνονται. Αν δει κανεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σε σχέση με τους πρώτους απολογισμούς και τις εκτιμήσεις που κάνει θα δει ότι ήδη σχεδόν συνομολογούμε ότι για το 2020 τους στόχους που έχουμε θέσει τόσο για την προώρη σχολική εγκατάλειψη όσο για, την, ε, για το ποσοστό των Ευρωπαίων που έχουν συμπληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και τα ποσοστά για την έρευνα φαίνεται ότι ήδη εκτιμάμε ότι δεν θα τα αγγίξουμε, ότι δεν θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Αν κανείς συνεκτιμήσει ότι στην ανακοίνωση αυτή της Επιτροπής δεν έχουμε κάποια εξειδίκευση σε ό,τι αφορά τους πόρους που αφιερώνουν τα κράτη-μέλη για την παιδεία, έχω την άποψη ότι εδώ ε, έχουμε μια σημαντική ευκαιρία και πρόκληση η Επιτροπή μας να τονίσει αυτά τα θέματα και ακριβώς να αναδείξουμε αυτό που είπε και ο εισηγητής, ότι προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους πρέπει να δίδουμε έμφαση, να λαμβάνουμε αποφάσεις πολιτικές τέτοιες που να τονίζουν ακριβώς αυτή την ανάγκη. Αν κανείς δει επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής και εγώ εισαγωγικά τοποθετούμε βεβαίως με τον εισηγητή θα έχουμε την ευκαιρία να ε, υποθέτω να ανταλλάξουμε πολλές φορές απόψεις ε, θα δει για παράδειγμα στις προτάσεις της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και μία πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την διανοητική ιδιοκτησία, ώστε αναγράφει η ανακοίνωση, ώστε να δοθεί έμφαση στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό το σε ότι αφορά την ανάπτυξη, όμως και εμεί ω Επιτροπή Παιδείας έχουμε σημαντικό ρόλο να επιτελέσουμε στα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό που τόσο τονίζουμε και βλέπουμε ότι τα προβλήματα την εποχή μας είναι πολύ σημαντικά. Ε, δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή των απόψεων. Ε, πραγματικά όμως και εγώ θέλω να συμφωνήσω ότι με αυτήν την διαδικασία που πλέον θα έχουμε για τα ε, εξάμεινα αυτά, για το ευρωπαϊκό εξάμεινο, θα μας δίνεται η ευκαιρία να είμαστε πιο κοντά στην σύνδεση των στόχων που έχουμε θέσει με τις πολιτικές που εφαρμόζονται και ας ελπίσουμε ότι και αυτό είναι κάτι που πρέπει να τονίζουμε και αυτό είναι θέμα όλων μας αλλά και της Προέδρου μας και της συνολικά του Κοινοβουλίου μας ότι αυτές οι, αυτές οι απόψεις που εκφράζουμε και καταθέτουμε και τελικά καταλήγουμε σε ένα κείμενο δεν είναι απλά μια θεωρητική προσέγγιση, είναι αποτελέσματα διαβούλευσης, πολύ μεγάλου προβληματισμού και τελικά ε, κρίσιμα συμπεράσματα για την επίτευξη των στόχων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υπενθυμίσω το εξή. Νομίζω ότι στην αρχή η ίδια η πρόεδρο μα είπε τι είναι το ευρωπαϊκό εξάμεινο, το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά πόσο άκουσα μέχρι, μέχρι τώρα. Το θέμα στο οποίο επέμεινε ο κύριος Τάκουλα είναι το θέμα της εγκατάλειψης του σχολείου. Άρα θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρόβλημα συντονισμού μεταξύ των πολιτικών των διαφόρων κρατών μελών. Διότι στη δεύτερη περίπτωση πρέπει να πω ότι υπάρχουν χώρες που μείωσαν πάρα πολύ σημαντικά τα κονδύλια τα οποία προορίζονται για την εκπαίδευση. Τι σημαίνει συντονισμός. Μπορούμε να κάνουμε συντονισμό μεταξύ μας. Η Κομισιό θα έπρεπε να το υπενθυμίσει αυτό, διότι η εγκατάλειψη του σχολείου δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει το παιδί το σχολείο. Πολλές φορές έχουμε σχολεία που εγκαταλείπουν στον δρόμο τα ίδια τα παιδιά. Γιατί? Διότι μειώθηκαν οι πόροι, μειώθηκαν οι εκπαιδευτικοί και ότι είναι 20 παιδιά στην τάξη υπάρχουν 40. Άρα μερικά μένουν στην άκρη. Ας μην ε, εθελοτυφλούμε λοιπόν. Υπάρχουν πολύ σημαντικά προβλήματα ε, σε κάποιες χώρες τις οποίες μειώθηκαν σημαντικά οι πόροι που δίδονται στην εκπαίδευση επαναλαμβάνω. Θα πρέπει να συντονιστούμε λοιπόν για να καταπολεμήσουμε τέτοιου είδους τάσεις. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Κώστα. Ναι. Και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Κύριε Τάκουλα, σωστά αναφέρατε προηγουμένως ότι ο στόχος του 10% για τη σχολική εγκατάλειψη είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Στο χώρα μου το ποσοστό αυτό είναι της τάξης 15-16%. Βεβαίως ξέρουμε ότι η Ευρώπη σήμερα παρτίζεται από πολύ διαφορετικές χώρες. Σωστά υπενθυμίσατε ότι 10% είναι η υποχρέωση για φέτος, σύμφωνα με τους στόχους της Λισαβόνας. Προηγουμένως είπε κάτι το πολύ σωστό συνάδελφος. Βεβαίως θα πρέπει να τηρήσουμε την αρχή της επικουρικότητας, αλλά έχουμε συγκριτικές μελέτες, συγκριτικές αναλύσεις, ξέρουμε τι γίνεται, γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα στι χώρες να μην μειώσουν τις επενδύσεις τους και τα κονδύλια του σε θέματα εκπαίδευση. Θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε στο έγγραφο αυτό σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τώρα, για να μην ε, έχουμε τις ίδιες απογοητεύσεις που είχαμε στα πλαίσια της Λισαβόνας, δεδομένου ότι υπάρχουν ανοιχτές αυτές ε, συγκρίσεις και μελέτες θα πρέπει να συντονιστούμε καλύτερα για να δούμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας για το 2020. Όταν μιλούμε για την εκπαίδευση δεν ε, λέμε καθόλου ότι θα πρέπει να κάνουμε επενδύσεις για να είναι πάντα ενημερωμένο το διδακτικό προσωπικό. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει οι διαδικασίες της Κοπενχάγης και της ε, Μπολόνια να ενισχυθούν και να υπάρχουν ίδιες δυνατότητες μεταξύ όλων των μαθητών και φοιτητών όσον αφορά την ισοδυναμία και την αναγνώριση των πανεπιστημιακών του πτυχίων. Νομίζω ότι πολλά, λοιπόν, πολλά μπορούμε να κάνουμε και πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό. Πρόκειται για δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να ενταχθούν στο κείμενο για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Πρέπει να συνηθίσουμε πρώτα την έκφραση. Ε, λίγο παράξενη ονομασία για αυτό που θέλουμε. Δεν ξέρω αν ακούγεται σε άλλες γλώσσες διαφορετικά. Γιατί μερικοί φαντάζονται ότι είναι πανεπιστημιακό εξάμεινο ή... Είναι περίεργο. Ε, είναι η χαρακτηριστική ευρωπαϊκή γλώσσα. Αν θέλουμε κάποια αποτελέσματα, αυτά ποια θα είναι. Έγκαιρα μέσα στο χρόνο θα βλέπουμε τι έχουν σχεδιάσει στον προϋπολογισμό τους τα κράτη-μέλη για τους διάφορους τομείς και θα πρέπει να ε, δείξουν τι κάνουν και στους άλλους, στους υπόλοιπους τομείς. Οι κυβερνήσεις ε, έχουν ε, υποσχεθεί πολλά να αυξήσουν τα ποσοστά των πολιτηριούχων δευτεροβάθμιας κλπ. Είναι πολλοί οι στόχοι, όχι όσο στη στρατηγική της Λισαβόνας που είχαμε βέβαια πάρα πολλούς στόχους, υπερβολικά πολλούς και δεν πραγματοποιήθηκε κανείς, γιατί δεν υπήρχε κανείς ο οποίος θα παρακολουθούσε το θέμα. Δηλαδή έγινε η δουλειά που έπρεπε. Κανείς δεν ρώτησε τους υπουργούς παλιά αν έκαναν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πρόβλημα. Γι' αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο αυτό θα κάνει. Θα υπάρχει δηλαδή απολογισμός. Έγινε η δουλειά. Και Οι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο μίλησαν για το πώς ε, θα μπορέσει να επιδράσει θετικά για να μην μείνουν επί χάρτου όλα αυτά, τα, ε, όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε, αλλά να βγει ένα ρεζουμέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για την Κομισιόν, η Κομισιόν πιστεύω ότι πρέπει να πάρει θέση εδώ σε αυτή τη προγραμματική περίοδο διαπιστώνουμε ότι η πολιτική πηγαίνει προς μία κατεύθυνση. Η πολιτική όμως πρέπει να αποσκοπεί στην ε, οικοδόμηση του μέλλοντος. Δεν πρέπει να μας απασχολεί δηλαδή η διαχείριση των τρεχουσών ε, καταστάσεων, αλλά πρέπει να δουλεύουμε με προσανατολισμό στο μέλλον. Και πρέπει να μάθουμε από αυτά που δεν λειτουργήσαν, δυστυχώς, όπως η ε, ατζέντα της Λισαβόνας. Ε, διάβασα κάποια έγγραφα της Κομισιόν και μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στερείται κάποιων βασικών γνώσεων και επιγνώσεων η Κομισιόν. Στη Φιλανδία, για παράδειγμα, λέμε συχνά ότι ίσως δεν χρειάζεται η γεωργία πια καθόλου γιατί θα πρέπει να αυξηθεί η επιχειρηματικότητα ή ε, ε, α, δεν χρειαζόμαστε ε, παραγωγή ενέργειας γιατί η ηλεκτρική ενέργεια βγαίνει από την πρίζα. Ε, χάνουμε δηλαδή κάποιες οριζόντιες διασυνδέσεις και ε, επαφές που είναι σημαντικές και ορισμένες ανάγκες θα καταγραφούν τώρα όπως ποιότητα στην εκπαίδευση, βιώσιμη ανάπτυξη βάση των, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού χρειάζεται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό χωρίς αυτό δεν υπάρχει ανάπτυξη, ανάπτυξη εξαρτώμεθα από το σύστημα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίως εξαρτώμεθα και από εξαιρετικούς, χρειαζόμαστε και εξαιρετικούς ε, καθηγητές. Άρα πρέπει να γίνει επένδυση και στη διαβίου και στην εκπαίδευση κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η στόχοι είναι καλή, αλλά όπως είπαμε, ένας στόχος είναι να ε, μηδενιστεί η εγκατάλειψη του σχολείου είναι πολύ φιλόδοξος στόχος, ε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον πετύχουμε, αλλά έτσι θα κινηθούμε προς την καινοτομία και την ε, θέμενη αξία στην Ευρώπη. Ωραία. Κλείνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση προς το παρόν και εξαντλήσαμε και το, την ημερήσια διάταξη αφού δεν μπόρεσε η κυρία ε, η Επίτροπος κυρία Βασιλείου να έρθει, λύεται συνεδρίαση, η Ευχαριστούμε τους διερμηνείς, θα παραμείνουν όμως για να συνεχίσουμε με τους συντονιστές. Όσοι δεν είναι συντονιστές και συνεργάτες μας παρακαλούνται να αποχωρήσουν.